Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διαταξή έγκριση αυτής. Βρίσκεται στους φακέλους σας. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνεται χωρίς τροποποίησης. Πρέπει να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Κατά πρώτον, η αυριανή συνεδρίαση 3ης 19 Μαρτίου το απόγευμα κατ' εξαίρεση θα ξεκινήσει στις 3.30. Σε κάθε περίπτωση θα αποσταλεί mail σε όλους τους συναδέλφους που είναι μέλη της Επιτροπής μας, ώστε να τους ενημερώσουμε θα ξεκινήσουμε στις 3.30 λοιπόν, διότι προηγουμένως υπάρχει η διάσκεψη των Προέδρων που είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Και θα διαρκέσει από τις 2.30 έως τις 3.30. Γι' αυτό και η δική μας συνεδρίαση Επιτροπής θα ξεκινήσει στις 3.30 και θα ολοκληρωθεί στις 7. Αυτά για αύριο, 3η 19 Μαρτίου. Επιπλέον, έχουμε μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Το σημείο 7 άλλαξε θέση και πήγε στη θέση του 19. Η έκθεση Τσίτσεστερ λοιπόν θα συζητηθεί αύριο 19 Μαρτίου μετά τις ψηφοφορίες. Ενώ η έκθεση Τόγια θα συζητηθεί 18 Μαρτίου το απόγευμα. Σήμερα, το σημείο 9 τελικά αναβάλλεται για τις συνεδρίες της 24ης 25ης Απριλίου. Θα το δούμε από κοινού με την εξέταση του σχεδίου έκθεσης του συναδέλφου Μπουτικόφερ για τον προπολογισμό του 2014 καθώς και την εντολή για τριμερή διάλογο. Στο σημείο 3 τώρα έχουμε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Φεβρουαρίου και αυτά βρίσκονται στους φακέλους σας. Οπότε και εδώ, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης κοινοτικό σύστημα καταχώρησης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών. Εισηγητής είναι ο κύριος Μπέλα Κόβατ, στον οποίο θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Και μετά θα ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές. Κύριε Κόβατ, για, πέντε λεπτά. Uh, Ευχαριστώ. 3 Φεβρουαρίου του 2012 αποφάσισε το Συμβούλιο να ζητήσει γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 7 της Ευρατόμ σχετικά με μια πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που καθορίζει ένα κοινοτικό σύστημα καταχώρησης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών. Οι διατάξεις έχουν ως στόχο την ε, ασφάλεια και των εργαζομένων αλλά και γενικότερα του κοινού. Η νομική βάση είναι το κεφάλαιο 3 της συνθήκης βάση της ε, Ευρατόμ και το άρθρο 31 και 32. Η πρόταση αυτή, πρόταση για κανονισμό, αντικαθιστά τις εθνικές διατάξεις και διαδικασίες προκειμένου να αναφέρονται οι μεταφορές ραδιενεργών υλικών και τις αντικαθιστά με ένα νέο σύστημα. Βασικά θα υπάρχει και απλοποίηση του γραφειοκρατικού άχθους και θα υπάρχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας από ραδιενεργά υλικά. Ως εισηγητής λοιπόν εξέτασα την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που φροντίζει να ε, γίνεται και καλύτερος έλεγχο των μεταφορών αυτών. Παρ' όλα αυτά έχω κάποιες βελτιώσεις στο κείμενο. Προκειμένου να υπάρχει ίση μεταχείριση των μεταφορέων, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να δίνουν το πιστοποιητικό κατοχώρησης και να υπάρξει και αναρμόνιση της διαδικασίας καταχώρησης. Και αυτό προκειμένου να μην υπάρχει περιττή γραφειοκρατία. Η εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονική υπογραφή. Το σύστημα καταχώρησης πρέπει να είναι ασφαλές, ισχυρό και να λειτουργεί πλήρως προτού να αρχίσει η ισχύ του κανονισμού. Και επίσης πρέπει να υπάρξει και ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, των εθνικών αρχών δηλαδή, και να υπάρξουν τα συστήματα καταχώρησης σε όλες τις χώρες μέλη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μεταφορές διασυνοριακά. Η μεθοδολογία επίσης πρέπει να είναι ίδια με εκείνη που ισχύει στι ισχύουσε τώρα οδηγίε. Οι ορισμοί, οι προδιαγραφές ιδιαίτερα αυτά που προτείνει η Διεθνής ε, Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας. Το θέμα της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, για παράδειγμα. Πρέπει για κάθε δραστηριότητα να ξέρουμε κατά πόσο εμπίπτουν στο εύρος εφαρμογής του συγκεκριμένου κανονισμού ή όχι. Ε, επίσης, να συμπεριλαμβάνονται προδιαγραφές ασφάλειας της οδηγίας Όπω επίσης και εκείνες που αναφέρονται και τα στοιχεία που αναφέρονται σε άλλε οδηγίε που έχουν να κάνουν με ιατρικά στοιχεία, με επίπεδα ραδιενέργειας, με διάφορες ε, δραστηριότητες, σφραγίσματος για παράδειγμα, ε, μεταφοράς ε, κοντέινερς που μεταφέρουν αδιανεργά υλικά κλπ. Πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση επίσης του ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών. Το θέμα της καταχώρησης είναι πολύ σημαντικό. Οι εθνικές αρχές πρέπει να έχουν όλα τα δεδομένα που χρειάζονται όσον αφορά την καταχώρηση αυτή, για να μην υπάρχει τίποτα πλαστό και να μπορούν να κάνουν τον έλεγχο σωστά. Δεν καλύπτονται εδώ οι μεταφορές ραδιενεργών δηλαδή, υλικών από αέρος ή διαθαλάσσεις. Πρέπει να υπάρξει ένα νέο σύστημα καταχώρησης για αυτές τις περιπτώσεις. Η διαθαλασσης πρεπει να υπαρξει ενα νεο Επιτροπή πρέπει να δει τι δυνατότητες υπάρχουν και τι συστήματα πρέπει να προτείνει από αυτά που ήδη υπάρχουν για αυτές τις περιπτώσεις. Κατά τη γνώμη μου, η πιο αποτελεσματική λύση είναι αυτή που προτείνουμε σήμερα γιατί μπορεί να εφαρμοστεί και γρήγορα. Παρόλο βέβαια που πρέπει να πούμε ότι ισχύουν διαφορετικά συστήματα στις μεταφορές διαέρος ραδιονεργών υλικών. Στόχος πάντως της σημερινής πρότασης είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να ενισχυθεί η διαφάνεια και να μειωθεί ο φόρτος των μεταφορέων, συγχρόνως βέβαια φροντίζοντας η ασφάλεια να είναι στο ανώτατο επίπεδο. Όσον αφορά τώρα τις επιπτώσεις του κανονισμού αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο χρόνια αφότου τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει να μας ενημερώσει με έκθεσή της για τις επιπτώσεις αυτές. Τέλος, πιστεύω ότι ο μεταφορέας θα πρέπει να ενημερώνει τα δικά του τα ε, στοιχεία από μόνος του, χωρίς να επιβάλλεται επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Κόβατς και τώρα ο συνάδελφος Κάριντς ο οποίο θα μιλήσει στη θέση του κυρίου Μαρινέσκου, που είναι ο σκιώδη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Μιλάω εκ μέρου του κυρίου Μαρινέσκου. Καλωσορίζω την ε, πρόταση αυτή, διότι ένα ευρωπαϊκό κεντρικό σύστημα για την καταχώρηση των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών για την ε, χερσαία μεταφορά είναι απαραίτητο. Όλοι οι πολίτε θα πρέπει να προστατεύονται από τι ιονίζουσε ακτινοβολίε. Το θέμα είναι κατά πόσον θα είναι ασφαλέ ένα τέτοιο ηλεκτρονικό σύστημα και ποιε εγγύσει θα υπάρχουν από του συμμετέχοντε τρίτων χωρών για του μεταφορεί που έρχονται δηλαδή στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συμμορφώνονται με τι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα συμβεί εάν το κάτω μέλο του οποίου επικράτεια θα είναι η πρώτη από την οποία θα διέλθει ένα μεταφορέα έχει δώσει κατά την άδεια για την καταχώρηση του μεταφορέα ραδιενεργού υλικού από τρίτη χώρα ή εάν αρνηθεί κάτι τέτοιο ή να αναγνωρίσει έναν επόμενο κράτος ε, την ε, άδεια του πρώτου κράτους διέλευση. Έπειτα, ποιε είναι εγγυήσει για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι εγκεκριμένοι μεταφορεί είναι απολύτως ασφαλεί και πλήρω μορφούνται, εφόσον προέρχονται από τρίτες χώρες, με τι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδρομή. Ιδίω επειδή μιλάμε για ραδιενεργά υλικά υψηλή ακτινοβολία ε, κάποιε φορέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Κουάντρας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή κανονισμού θέτει έναν στόχο τον οποίο πάντα πρότεινε στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ασφάλειας και να τηρούνται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ακούσαμε, θέλουμε να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρηση μεταφορέων ραδιενεργών υλικών, προκειμένου να γνωρίζουμε πόσοι είναι, με τι ακριβώς ασχολούνται και τι μέτρα ασφάλειας εφαρμόζουν. Συγχρόνως, τα κράτη-μέλη θα μπορούν πιο εύκολα να ελέγχουν τις προδιαγραφές ασφάλειας στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών, προκειμένου να μπορούν έτσι να προστατεύουν και τους επαγγελματίες, αλλά και γενικά τον κόσμο που κινδυνεύει να εκτεθεί σε τέτοια ραδιενέργεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι μεταφορείς. Γιατί, γιατί τώρα επικρατούν διαφορετικά συστήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμφέρει να έχουν ένα ενιαίο σύστημα. Αν υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα καταχώρησης, θα υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερο κόστος, άρα θα είναι πολύ καλό για το τομέα αυτόν και οικονομικά. Τώρα, συγχρόνως, πρέπει να καταργηθούν τα εθνικά συστήματα καταχώρησης εφόσον θα έχουμε ένα νέο ευρωπαϊκό. Δεν πρέπει να προσθέσουμε ένα ακόμα γραφειοκρατικό επίπεδο. Όχι, πρέπει να το αντικαταστήσουμε. Τώρα σε σχέση με τα κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρεί κανείς για να πάρει την άδεια και να μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα αυτό. Από αυτό που ξέρουμε από την Ευρατόμ το 96 κάθετος 29 για την προστασία των εργαζόμενων και του κοινού από τη ραδιενέργεια. Υπάρχει λοιπόν αυτή και υπάρχει και οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αναφέρεται στις επικίνδυνες ουσίες. Πρόκειται για οδηγίες και οι εφαρμοστικές πράξεις βάζουν κάποιες προϋποθέσεις πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες μερικές φορές μεταξύ τους αποκλίνουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Δίχως άλλο, ο συγκητής θα το λάβει υπόψη του αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο ο κύριος Τζόρνταν. Κυρία Τζόρνταν. Ε, Σας ευχαριστώ, Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος προετοίμασα μία γνωμοδότηση και πρέπει να σας πω ότι και στις δύο επιτροπές θα προασπίσω την ίδια γνώμη. Θεωρώ ότι είναι καλή η πρόταση αυτή για το σύστημα καταχώρησης και πέρα από αυτά που ήδη είπαν οι συνάδελφοι για την βελτιωμένη ασφάλεια και ούτω καθεξής, συνεπάγεται μεταξύ, άλλος, μεταξύ άλλων και λιγότερη γραφειοκρατία για τους μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό. Καταργούνται εμπόδια τα οποία προκύπτουν στην παρούσα φάση από, τα διαφορετικά, από τις διαφορετικές νομοθεσίες. Υπάρχει λοιπόν αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων αυτών, αλλά αυτό θα γίνει μόνο εφόσον υπάρχουν ενιαία πρότυπα. τάλα στο σύστημα αυτό θα μπορούσε να καταστεί επιζήμιο, γιατί δεν θα ήταν αξιόπιστο. Και αυτό θα προκαλούσε φυσικά μεγάλη δυσπιστία από πλευρά των πολιτών. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή που έχουμε μπροστά μας. Όταν δεν πληρούνται οι απαραίτητες ε, προδιαγραφές θα πρέπει να τίθενται, να επιβάλλονται μέτρα από τις αρχές προκειμένου ο εκάστοτε μεταφορέας να αναγκάζεται να προβαίνει σε αλλαγέ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η δραστηριοποίηση, η μεταφορά από τον μεταφορέα αυτόν μέχρι ότου διορθωθούν τα ελαττώματα. κάποια διοικητικά όργανα ενδεχομένως να είναι πιο αδύναμα από ό,τι άλλα και ενδεχομένως να προκύψουν σπάλματα. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να έχουμε προβλέψει για τέτοιες περιπτώσεις. Θα πρέπει να ορίζονται σαφώς οι προθεσμίες. Προθεσμίες για το πότε θα πρέπει να αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο τα περί για παράδειγμα. Και έχω και κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση, αυτό το σύστημα θα πρέπει να ισχύει για όλες τις πηγές ραδινεργών υλικών και ραδινεργής ακτινοβολίας, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, μάλλον κανονικά εξαιρούνται οι στρατιωτικές χρήσεις. Κάτι άλλο. Πόσο θα κοστίσει το σύστημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας αγγιηθεί ότι δεν θα συμβεί σε άλλες περιπτώσεις όπου οι τιμές δημορφώθηκαν πολύ χαμηλές. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Θα πάρει κάποιος το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την θετική σας στάση ως προς την πρότασή μας. Οι βασικές, η οδηγία για τις βασικές προδιαγραφές ασφαλείας βάσει της συνθήκης Euratom καθορίζουν βασικές προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού σε ό,τι αφορά τις ιονίζουσες ακτινοβολίες. Καθορίζει όλες τις πρακτικές που ενέχουν κίνδυνο και επιρροή από ιονίζουσες ακτινοβολίες και βάσει της οδηγίας αυτής οι μεταφορές υπόκεινται σε υποχρέωση υποβολής έκθεσης και διαδικασία διοδότησης. Η πρότασή μας υποκαθιστά το σύστημα υποβολής εκθέσεων και αδειοδότησης στα κράτη-μέλη, προκειμένου να ισχύουν βασικές προδιαγραφές ασφαλείας, αλλά με ενιαίο σύστημα καταχώρηση που να ισχύει με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Με τέτοια μετατροπή θα απλουστευτούν οι διαδικασίες, κάτι που υπόθηκε ήδη, θα περιοριστεί το διοικητικό άχθος για τους μεταφορείς και θα εξαλειφθούν οι φραγμοί εισόδου το καθοριστικό στοιχείο της προτινόμενης νομοθετικής έκθεσης είναι το ηλεκτρονικό σύστημα για την καταχώρηση των μεταφορέων. Υπάρχουν εδώ κάποιες ερωτήσεις από ό,τι άκουσα. Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατόν το σύστημα να λειτουργήσει πρωτοεγκριθεί εγκριθεί ο κανονισμός. Υπάρχει και μια δημοσιονομική διαδικασία και τα κονδύλια μπορούν να δαπανηθούν αυτή τη στιγμή εγκριθεί ο κανονισμός. Για να καταλάβετε λίγο το κόστος που μας αφορά εδώ, έχουμε να κάνουμε με ένα εκατομμύριο ευρώ περίπου. Οπότε οι ειδικοί μας, οι εμπειρογνώμονες, ε, της οι ειδικοί της πληροφορικής, θα κοιτάξουν να υπάρχει ένα σύστημα πολύ ασφαλές για την ηλεκτρονική καταχώρηση. Ο κανονισμός προβλέπει μια σταδιακή ε, υλοποίηση και θα ισχύει για κάθε μεταφορέα που μεταφέρει ραδιονεργά υλικά εντός κοινότητας ή με προέλευση από τρίτη χώρα προς την κοινότητα. Προφανώς οι αιτήσει μεταφορέων τρίτων χωρών θα εξετάζονται εξίσου εξονυχιστικά με, το, με αυτές των μεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα ισχύει όμως για μεταφορείς που μεταφέρουν ε, ραδιενεργά υλικά αεροπορικός ή διαθαλάσσης. Αυτό νομίζω ούτως ή άλλως αναφέρθηκε. και νομίζω ότι έχουμε ήδη ένα προηγμένο σύστημα, αρκετά εξελιγμένο για αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, <clears throat> για τις πτυχές της ασφάλειας, ήδη υπάρχει νομοθεσία σχετική, ο κανονισμός δηλαδή του Συμβουλίου για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών μεταξύ κρατών μελών, καθώς και ο κανονισμός του Συμβουλίου για την επίβλεψη και τον έλεγχο των ραδιενεργών υλικών και καταλήπων καυσίμων. Οι κανονισμοί αυτοί θα συνεχίσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται. Αυτά τα νομοθετικά, αυτά τα νομοθετήματα σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ασφαλή ε, προστατευμένη και ελεγχόμενη μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί ρώτησαν για το και τα κοινά ή εναρμονισμένα κριτήρια καταχώρησης. Το θέμα αυτό συζητιέται και στο Συμβούλιο, στην αρμόδια ομάδα εργασίας, την ομάδα για την ατομική ενέργεια, βρίσκεται σε εξέλιξη και αποκινούμε τα κράτη-μέλη. Σκεφτόμαστε ακριβώς ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση. Είμαστε ευγνώμονες προς τον εισηγητή σας που ανέφερε ως μια από τις πρώτες προτεραιότητες την ε, κατάρτιση κριτηρίων για την καταχώρηση. Κυρία Πρόεδρε, για πιο συγκεκριμένα ζητήματα, ευχαρίστως θα δώσουμε απαντήσεις στον εισηγητή βάσει των όσων πληροφοριών έχουμε συγκεντρώσει από τα κράτη-μέλη και προφανώς με τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να αποφύγουμε στρεβλώσεις ανταγωνισμού στο σύστημα. Πιστεύω όμως ότι ο απότερος στόχος αξίζει τον κόπο να τον επιδιώξουμε προκειμένου να έχουμε έναν εναρμονισμένο, μοναδικό και ενιαίο σύστημα καταχώρησης που να επιτρέπει στους μεταφορείς μας να συνεχίσουν τις διασυνοριακές μεταφορές ραδιενεργών υλικών ώστε οι μεταφορέ να παραμένουν ασφαλείς για να μην πω ασφαλέστερε από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο λόγο στον συνάδελφο Κόβατ για τα συμπεράσματά του. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να δούμε ποια είναι τα κοινά σημεία τα οποία τελικά να μπορούν να αποδεχτούν τα κράτη-μέλη και τα οποία να μπορεί να δεχτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίε και κύριοι, αυτό που σας ζητάω είναι να μου στείλετε ό,τι σχόλια έχετε με λεπτομέρειες και ό,τι τροπολογίες έχετε επίσης να τις υποβάλλετε και εγώ να ξέρετε ότι θα τις λάβω υπόψη μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Κόβατ. Να θυμίσω τις προθεσμίες. Εξέταση της έκθεσης 13 Μαΐου 16 Μαΐου το μεσημέρι λίγη η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και Νομίζουμε θα μπορούμε να ψηφίσουμε στις 19-20 Ιουνίου και να περάσει στην Ολομέλεια τον Ιούλιο η έκθεση. Και τώρα, έκθεση Κάρινς. Συγκεκριμένα δύο εκθέσεις. Θα τις δούμε ταυτόχρονα. Σημεία 5 και 6. Οπότε έχουμε το διπλάσιο χρόνο και θα δώσουμε και διπλάσιο χρόνο, κύριε Κάριν, σε εσά για την πρώτη σα παρέμβαση. Έχετε το λόγο. Σημεία 5 και 6. Συμφωνήσαμε να τα δούμε από κοινού. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο σε ό,τι αφορά τον περιοδικό έλεγχο των χαρακτηριτών οχημάτων. Φαίνεται ότι αυτό είναι αρκετά ε, έντονο θέμα, μάλλον ε, θέμα που προκαλεί έντονα συναισθήματα, αν και όχι τόσο για την Επιτροπή μας. Γνώρισα πολλά καινούργια άτομα που μου απορουσίασαν πολλά καινούργια αριθμητικά στοιχεία και καταλαβαίνω πλέον ότι πάντα για κάθε θέμα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που το υποστηρίζουν και που αντιτίθενται είναι λοιπόν αρκετά περίπλοκο το θέμα. Στην έκθεσή μου έχω συμπεριλάβει κάποιες σχετικές ε, τροπολογίε Το θέμα καταρχάς του πόσο συχνά θα πρέπει να επιθεωρείται ένα όχημα και κατά πόσον το θέμα των πόσων χιλιόμετρων ε, τι υπέρβαση υπάρχει. Αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και ιδιαίτερα για τους Βρετανούς αγρότες, αλλά νομίζω ότι βασικά είναι ένα θέμα που αφορά την Επιτροπή Μεταφορών. Πρόκειται για ένα θέμα α, ερμηνείας των στατιστικών στοιχείων που έχουμε ακούσει ο καθένας. Εγώ επικεντρώνομαι πιο πολύ στα θέματα εκείνα τα οποία που θεωρώ ότι θα εξυπηρετήσουν το κοινό συμφέρον. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα στοιχεία του χιλιομετρητή, τα οποία συχνά υπόκειται νοθεία, φαίνεται. Και τελικά συχνά ε, δεν είναι ακριβή τα στοιχεία αυτά. Αν υπήρχε όμως ένας ηλεκτρονικός έλεγχος των στοιχείων αυτών, αυτό σίγουρα θα διευκόλυνε τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με θέματα ασφάλειας. το πόσα χιλιόμετρα έχει ένα όχημα ε, σχετίζεται και με την ασφάλειά του σε ό,τι αφορά την έκθεση για την περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Το θέμα είναι ο μετρητής λοιπόν των διανυθέντων χιλιόμετρων. Θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και αυτό το αποτυπώνω σε διάφορες ε, ε, τραπολογίες. Για το άλλο, την άλλη έκθεση τώρα, σε ό,τι αφορά το τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματική χρήσεω. Το να σταματάμε, για παράδειγμα, ένα φορτηγό στο δρόμο για να ελέγξουμε αν πληρεί τι προδιαγραφέ. Μία μεγάλη δυσκολία είναι ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πρότυπα μεταξύ των κρατών μελών. Μεταξύ άλλων και τα θέματα τεχνικής επιθεώρησης. Άρα, εξαρτάται αν το όχημα ελέγχεται στο χ ή ψ κράτο μέλο ένα όχημα το οποίο περνάει τον έλεγχο σε ένα κρατός μέλος μπορεί να μην το περνούσε σε κάποιο άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση από τεχνικής άποψης. Να θεωρούταν δηλαδή ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Χρειαζόμαστε λοιπόν με έναν τρόπο να προάγουμε μια κοινή ερμηνεία του τι είναι ασφαλές και τι είναι μη ασφαλές. Στα κράτη-μέλη ε, η κατάσταση είναι διαφορετική και σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά οχήματα και πολλές χώρες που είναι χώρες διαμετακόμισης. Α, γι' αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις χώρες αυτές. Άλλε πάλι χώρες είναι στην περιφέρεια της Ευρώπης. Ίσως λοιπόν για αυτές να μην είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό, μιας και δεν περνάνε από αυτές τα οχήματα που προορίζονται για μια άλλη χώρα. Στην Ευρώπη σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων με ηλεκτρονικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει οι οδηγοί να έχουν τις πιστοποιήσεις, τις άδειε στο χέρι τους. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να διατίθενται ηλεκτρονικά. Και όσο πιο πολύ συμμετέχουν τα κράτη-μέλη στο σύστημα αυτό, τόσο μεγαλύτερη και καλύτερη θα είναι η βάση για την ε, διατύπωση κοινών προτύπων. Θεωρώ ότι και αυτό αποτελεί ένα στόχο στο πεδίο εφαρμογή των προτάσεων αυτών. Και φυσικά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση βάσει της χώρας προέλευσης σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των ελέγχων αυτών. Επίσης, προτείνω κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά τι, το γίνεται, τι γίνεται όταν ένας επιθεωρητής, ο οποίος έχει σταματήσει ένα όχημα, διαπιστώσει σοβαρές αδυναμίες, σοβαρά αλατώματα. Κάτι το οποίο αποτελεί προφανή και άμεσο κίνδυνο. Είτε για τον οδηγό, είτε και για οποιονδήποτε άλλο φυσικά στον δρόμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει λίγο πολύ να έχει ο επιθεωρητής το δικαίωμα να διασφαλίσει ότι το όχημα θα πρέπει να ε, καταστεί ασφαλές. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο άμεσοι. Ο επιθεωρητής θα πρέπει να έχει την υποχρέωση να μεταβεί το όχημα αυτό στο πιο κοντινό γκαράζ προκειμένου να καταστεί ασφαλές. Έχω, κατα... Έχω υποβάλει μια σχετική τροπολογία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό, αλλά ίσως όχι απαραίτητα από την πλευρά της Επιτροπής Βιομηχανίας. Άρα, τονίζω, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Όσο πιο πολύ, τόσο καλύτερα. Όσο πιο πολύ συμμετάσχουν στο σύστημα αυτό. Τόσο πιο ασφαλές θα είναι το σύστημα ταφρών στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκλάντε τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Κάριντς. Θα ήθελα εξ ονόματο του κυρίου Λάνε, που δυστυχώς δεν μπορεί να παραβρεθεί εδώ σήμερα, να σας πω ποια είναι η άποψή του. Αυτός, αυτή η πρόταση, πέρα από το, τις οδικές μεταφορές, επηρεάζει και την βιομηχανία σε ό,τι αφορά το σημείο 5 για τα φορτηγά μα. Άρασαν ε, οι τροπολογίες 5, 6 και 7 τροπολογία 6 για να είναι πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος. Ε, πρέπει να χρησιμοποιούνται ιστορικά δεδομένα για την τροπολογία 7. Λογικό είναι αυτό σε ό,τι αφορά τις δεσυνοριακές πωλήσει, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν ίδια στάνταρ, τα ίδια πρότυπα. Θα πρέπει να σκεφτούμε τέτοιες προσθήκες για το 3-7 για τον ορισμό των ιστορικών οχημάτων. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ακριβείς ε, στη διατύπωσή μας. Τα ιστορικά οχήματα συνήθως ε, είναι πιο φροντισμένα από τα απλά παλιά αυτοκίνητα και είναι μεγάλη η αγορά στην Ευρώπη με 25 δισεκατομμύρια ε, κύκλο εργασιών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σαφή ορισμό. και είναι οι νομοθεσίε που ισχύουν στα διάφορα κρατημέλα στο άρθρο 3 σημείο 9 για τον ορισμό των περιοδικών τεχνικών ελέγχων. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ακριβεί, θεωρώ στο 4-3. σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στι πληροφορίε για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για κατασκευαστέ και για τα α, γκαράζ. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ε, δυνατότητες όπως το onboard diagnose για να είναι δίκαιος ο ανταγωνισμός. Στο 5-2 τώρα, δεδομένων ε, των ε, προδιαγραφών για τα οχήματα και δεδομένη ε, των τεχνικών δυνατοτήτων που αναφέρετε και εσείς για την χειραγώγηση ενός χιλιομετρητή θα πρέπει να διαγραφεί η αναφορά στα χιλιόμετρα. Στο 6-2. θα πρέπει να είναι σαφές ότι θα πρέπει στον περιοδικό και εθνικό έλεγχο να ελέγχεται και ο τρόπος ε, καταχώρησης και ελέγχου όλων των ζητημάτων. Και μόνο σε περίπτωση που εντοπίζονται τέτοιες ε, τέτοια ασφάλματα, τέτοια σαλωτήματα, θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση. Στο 12.1 είναι καλός που για πρώτη φορά τίθενται ε, προδιαγραφές ποιότητας για τους ελεγκτές και τους επιθεωρητές, αλλά θα πρέπει τα κρατημέλη που έχουν ορίσει πιο υψηλά πρότυπα να έχουν δικαίωμα να συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα αυτό σε ό,τι αφορά τι ε, προδιαγραφέ αυτέ, Θα πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη κατάρτιστη. Με το 12.4 για τη συγκρισιμότητα των περιοδικών τεχνικών ελέγχων θα πρέπει να υπάρχουν τα ίδια πρότυπα πιστοποίηση, για παράδειγμα το ISO. Στο 15.1 η πρόσβαση στο, σε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να είναι δυνατή ε, για όλους τους φορείς και για το άρθρο 18 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας αυτή στην Ευρώπη. Μία μικρή παρατήρηση για το παράρτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κανόνες για τα αέρια, πολύ αυστηρούς. Θα πρέπει λοιπόν η έλεγχη να είναι ακριβείς προκειμένου να μην τίθεται θέμα αξιοπιστίας και για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο του καθαρού αέρα. Και εδώ θα πρέπει να κοιτάξουμε τις προτινόμενες επιθεωρήσεις για το τελευταίο θέμα για τα έξι, για τα γεωταχή θα πρέπει να κοιτάξουμε. Κάποια θέματα ισχύουν με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τα φορτίγα. Και κατά τα άλλα θεωρώ ότι ο κύριος Λάνε συμφωνεί με αυτά που προτείνεται και το θέμα της ε, ασφάλειας των χωρών διαμετακόμισης μεταξύ των οποίων συγκαταλέγει και η Γερμανία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Γκλάντε. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι... Θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα σε πολλά θέματα. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτά που προτείνει. Τα... Μας, βρίσκουν σύμφωνο αυτά που αναφέρονται, αλλά θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή Βιομηχανίας δεν θα πρέπει να απόσχει από την γνωμοδότησή της και από την εξέταση ζητημάτων τα οποία θα έπρεπε να συζητηθούν στην Επιτροπή Μεταφορών. Νομίζω ότι είναι σωστό να ακολουθήσουμε τον στόχο της ε, βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Θέλουμε ωστόσο τα προτινόμενα μέτρα να είναι αναλογικά με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και θεωρώ ότι η Επιτροπή Βιομηχανίας ε, πολύ καλά θα κάνει να γνωμοδοτήσει. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα παλιά οχήματα που πρέπει να περνούν από περιοδικούς ελέγχους κάθε χρόνο, να σας πω για τη χώρα μου ότι αυτό το εξετάσαμε ως δυνατότητα και ως σήμερα δεν έχουμε καταλήξει σε οριστικά επιστημονικά στοιχεία για την έκταση κατά την οποία θα συνέβαλε κάτι τέτοιο στη μεγαλύτερη δική ασφάλεια τουλάχιστον στην δική μου χώρα τα πράγματα είναι έτσι. Δεν φαντάζομαι αυτό να είναι διαφορετικό πολύ σε άλλες χώρες. 1% μόνο προκαλείται ατυχημάτων προκαλούνται από τα οχήματα αυτά. Μήπως λοιπόν ε, προκαλέσουμε ίσα ίσα μεγαλύτερη γραφειοκρατία σε περίπτωση που επιβάλλουμε τόσο μεγαλύτερου τεχνικούς ελέγχου. Να υποστηρίξω τώρα τα θέματα περί πρόσβασης ε, στα δεδομένα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα ελέγχου. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση και συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκλάντε ότι θα πρέπει το θέμα να είναι η λειτουργική ασφάλεια του οχήματο. Αυτό θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Θα πρέπει να τον ισχύσουμε στην έκθεση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα και να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι το οδικό δίκαιο είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και θα πρέπει λοιπόν να διευκρινίσω ότι δεν μπορούμε εδώ πέρα σε μια γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λέμε πότε θα πρέπει να σταματήσει να επιθεωρητή σε ένα όχημα και τι θα πρέπει να κάνει με το όχημα αυτό. Για παράδειγμα, αν ε, ένας ε, οδηγό από μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης έρθει με ένα φορτηγό το οποίο δεν πληρεί κατά τις σύγχρονες προδιαγραφές ε, από τη χώρα μου, θα το κάνει μόνο μια φορά γιατί είναι πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές που ισχύουν. Θεωρώ λοιπόν ότι η αγορά λειτουργεί με τρόπο που καθαρίζει τον δρόμο. Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω για την οδική ασφάλεια Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα διεύρυνση της νομοθεσίας για τις μηχανές. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε το κατά πόσον η τεχνική ασφάλεια και η τεχνική, η τεχνική λειτουργικότητα ε, μειώνουν τον κίνδυνο των ατυχημάτων, αλλά θεωρώ ότι χρειάζονται σε πρώτη φάση επιστημονικές έρευνες για το κατά πόσον είναι απαραίτητο να καταστούν υποχρεωτικές αυτές οι ρυθμίσεις για τον τεχνικό έλεγχο ή μήπως θα μπορούσε ενδεχομένως με τον τρόπο αυτό να προκληθεί μεγαλύτερη γραφειοκρατία και να μην βελτιωθεί απαραίτητα η οδική ασφάλεια. Υποστηρίζω λοιπόν την έκθεση σε κάθε περίπτωση, θα υποβάλω κάποιες συμπληρωματικές ε, τροπολογίες οι οποίες όμως δεν αντιτίθεται με το πνεύμα της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι τελικά θα είναι πολύ χρήσιμη και ε, καλή αυτή η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κράμερ. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ καταρχάς τον εισηγητή για την ε, συνεισφορά του. Θέλω να τονίσω ωστόσο ότι θα πρέπει να ελέγχουμε σε κάθε περίπτωση το τι γίνεται με τα ρημουλκούμενα οχήματα στην περίπτωση φρεναρίσματος. Το κατά πόσον δηλαδή υπάρχει σταθερότητα στο σύνολο οχήματος ρημουλκούμενου. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί σήμανση για το έμπροστρεν τμήμα του μέρους του οχήματος που ρημουλκεί, ώστε να υπάρχει προειδοποίηση ότι πίσω ακολουθεί το ρημουλκούμενο. Τα συγκεκριμένα λοιπόν όρια ταχύτητας που θα που θα ισχύουν για τα ρημουλκούμενα, εφόσον υπάρχει ρημουλκό, να μπορούν όντω να υλοποιούνται. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον κύριο Πρόντι. Ο κύριος Ανά. Ευχαριστώ. Είναι μια έκθεση που πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα. Τα περιλαμβάνει και δεδομένα πολύ σημαντικά. Ένα, ο τεχνικός έλεγχος πρέπει να παραμείνει ε, είτε μέσω πληροφορικής, είτε σε χαρτί, πρέπει να ισχύουν. Ένα αυτοκίνητο το οποίο πολλές φορές έχει ελεγχθεί, μερικές φορές αλλιώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα πραγματικά δεδομένα. Τώρα, όταν αλλάζουν κάποια ανταλλακτικά που είναι πολύ σημαντικά για την ασφάλεια του οχήματος, γνωρίζετε ότι τα ανταλλακτικά μερικές φορές είναι παραπημένα, είναι πλαστά, κάτι το οποίο αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Συνεπώς, τα ανταλλακτικά τα οποία αλλάζονται και το οποίο είναι σημαντικά για την ασφάλεια πρέπει να αναφέρονται κάθε φορά στον ε, τεχνικό έλεγχο. Επίσης, είναι απαραίτητο να ε, κρατήσουμε μεγάλες και σοβαρές κυρώσεις για εκείνους οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν λαθρεμπόριο με τα ανταλλακτικά. Δεν λέω ότι όλα διορθώνονται έτσι, αλλά αυτοί οι οποίοι ε, κάνουν κόλπα πρέπει να ξέρουν ότι οι κυρώσεις θα είναι πάρα πολύ βαριές. Θέλω να σταθούμε και σε δύο πράγματα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Το ένα είναι νομική πτυχή. Λέει ότι κάθε ιδιοκτήτη πρέπει να φροντίζει να είναι σε καλή κατάσταση το όχημα με το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο εκμεταλλεύεται τέλο πάντων. Είναι υπεύθυνο για την τεχνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το όχημα Εγώ ζω απέναντι από την Αγγλία, κάπου κοντά στο Καλέ. Κάπου ένα εκατομμύριο βαρεοχήματα περνάνε κάθε τόσο. Μερικές φορές αναγκάζονται να μείνουν στο Καλέ γιατί δεν είναι εντάξει το όχημά τους. Όταν όμως αυτό το λένε στον εργοδότη τους, τότε χάνουν τη δουλειά τους. Για τον εργοδότη τους λέει όχι πρέπει να κυκλοφορείτε. Ο κύριο υπεύθυνο λοιπόν για την μη καλή συντήρηση του οχήματο είναι ο ιδιοκτήτη, αυτός ο οποίο οργανώνει τη δουλειά. Ο οδηγό δεν μπορεί να μπαίνει αυτός πρώτα απ' όλα μπροστά στι ευθύνε του. Ο ιδιοκτήτη του οχήματο πρώτα απ' όλα είναι υπεύθυνο. Και κάτι ακόμα. για τις διακρίσεις εξαιτίας της πρόλευσης, καταγωγής της εθνικότητας. Εδώ θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τον κόπο να πάει λίγο στο καλέ και να δει τα φορτηγά που μας έρχονται είτε με πλοίο είτε από το τούνελ κάτω από τη μάχη. Θα διαπιστώσετε ποια είναι τα οχήματα τα οποία είναι σε καλή κατάσταση και ποια δεν είναι. Δεν θα σας πω εγώ ποια είναι η προέλευσή τους, αλλά αξίζει τον κόπο να πάτε επί τόπου να το δείτε με τα ίδια σας τα μάτια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλετε να παρέμβετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτή την ευκαιρία. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή σας και ιδιαίτερος στον εισηγητή σας. Εντυπωσιακή η δουλειά που έχετε κάνει για αυτό το τεχνικότατο και κάποιες φορές και έντονα συναισθηματικό θέμα. Καλά κάνατε όμως και τα αντιμετωπίσατε με τρόπο ουδέτερο και αντικειμενικό, προσθέτοντας στοιχεία που όντως χαρακτηριστικά προσφέρουν προστιθέμενη αξία και αρμόζουν σε μια επιτροπή υπεύθυνη για τα βιομηχανίας. Γενικώ μπορούμε να στηρίξουμε το σύνολο των τροπολογιών που προτείνει ο εισηγητή σα, διότι το αξίζουν σε κάποιες όμως περιπτώσεις και δεδομένου του βάρους που αναποθέτει ο συγητής σας στην αποτελεσματικότητα των εργαλείων πληροφορικής, εδώ θα έλεγα να επιδείξουμε μεγαλύτερη σύνεση, όπως για κάποιες συγκεκριμένε πτυχές. Λόγω χάρη χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριών, πλατφόρμα μεταξύ κρατών μελών, αυτή δεν έχει λειτουργήσει ακόμα πλήρως, οπότε πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποια σημεία που αναφέρονται και στο κείμενο ακόμα δεν έχουν επιτευχθεί. Συνολικά όμως μπορούμε να στηρίξουμε το σύνολο των προτάσεων για τις παρατηρήσεις που έγιναν ε, στην συζήτηση μόλις τώρα. Πράγματι, πρέπει να εργαστούμε εντατικότερα για τον ορισμό των ιστορικών οχημάτων. Το γνωρίζουμε αυτό. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Συνεργαζόμαστε στενά και με τους συναδέλφους σας της Επιτροπής Μεταφορών για τα επαγγελματικά προσόντα των επιθεωρητών κάποιοι βουλευτές ε, είπαν ότι θα έπρεπε να ενισχυθούν τα κριτήρια αυτά με τη συμπερίληψη λόγου χάρη συστάσεων συγκεκριμένου επίπεδου προδιαγραφών τη ΆΙΖΟ λόγου χάρη της ΆΙΖΟΕΛ. Αυτές είναι προτάσεις που μας βρίσκουν σύμφωνους για την περαιτέρω ενδυνάμωση των ευθυνών του ιδιοκτήτη, το ανέφερε ο κύριος ε, ένα από το καλέ. Ναι, είναι σωστό αυτό, αλλά μπορεί να δυσκολέψει κάποιο το πράγμα εάν θελήσουμε να το ενισχύσουμε. Και ακριβώς ε, συσχετιζόμενο με αυτό το σημείο είναι ότι θα ήθελε ο εισηγητής σας να αναγνωρίσει ότι στο πεδίο της εξαπάτησης με τον χιλιομετρητή θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ποινικά πρόστιμα, ποινικές κυρώσεις προβλέπονται ήδη. Χωρίς να θέλουμε λοιπόν να αποδυναμώσουμε το κείμενο, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας. Έντονη γλώσσα θα χρησιμοποιηθεί, καθώς αυτό είναι ένα από τα πολλά στοιχεία που προκαλούν κινδύνους για τα οχήματα που κυκλοφορούν στους οδούς της Ευρώπης. Και έπειτα δύο ακόμη σημεία που αναφέρθηκαν από βουλευτέ σα, Έχουμε να σχολιάσουμε ότι σε δύο σημεία η Επιτροπή στόχο δεν έχει να ε, κάνει πιο περίπλοκο το κείμενο, απλώς πρέπει να υπάρχουν αποδεκτικά στοιχεία και υπάρχουν ήδη πολλά τέτοια, ότι τα οχήματα είναι πηγή ατυχημάτων. Υπάρχει πραγματικά λόγος συγκεκριμένος, αναλογία και μάλιστα πολλαπλασιαστικά αυξάνεται ανάλογα με, την, με το πέρας της ηλικία των οχηματων Έξι, επτά έτη ηλικίας πολλές φορές βλέπουμε να προκαλούνται προβλήματα από αυτά. Θα πρέπει λοιπόν τουλάχιστον ετησίως τα οχήματα, ιδίως μεγάλης ηλικία, να υποβάλλονται σε έλεγχο. Και αυτό και για τα μοτοποδήλατα. Εφόσον αυτά γίνονται όλο και πιο περίπλοκα ως οχήματα, χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογικά μέσα σε σχέση με τα παλιότερα. Εδώ αυτό τα τα στοιχεία που έχουμε κρατήσει για να μελετήσουμε το συσχετισμό με τα ατυχήματα αποδεικνύουν ότι ετήσιος έλεγχος χρειάζεται και εκεί. Και αυτό για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια προς συμφέρον όλων. Κλείνω την εισήγησή μου λέγοντας ότι από εμά υπάρχει πλήρη στήληξη και οι τροπολογίες που προτείνονται νομίζουμε ότι θα βελτιώσουν αισθητά το κείμενο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριο Κάρνη για τα συμπεράσματά του. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλια που κάνατε και προσβλέπω στις ε, τροπολογίες σας. Δεν μου φαίνεται ότι απέχουμε πολύ. Και ίσως το θέμα να μην είναι τόσο πολιτικό μεταξύ των ομάδων. Ίσως να εξαρτάται πιο πολύ από τα κράτη-μέλη. Είναι καλό το μήνυμα. Είναι καλή η ένδειξη αυτή. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετά δυναμική η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Έχω κάποια σχόλια να κάνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, μας επεσήμανε τον κίνδυνο σε ό,τι αφορά μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγή ε, δεδομένα μεταξύ κρατών μελών. Εγώ πιστεύω ότι ακριβώς επειδή δεν δουλεύει το σύστημα αυτό, θα πρέπει να το τονίσουμε στην έκθεση. Αν δεν υπάρχει πίεση από πλευρά Κοινοβουλίου, από πού θα υπάρξει πίεση. Είναι σημαντικό στοιχείο λοιπόν και θα ήθελα να αντιτηρηθεί στην έκθεση. Ένα άλλο σχόλιο σε ό,τι αφορά τις νομικές κυρώσεις. Ε, Τροπολογία 9, άρθρο 9, παράγραφος 2. Στον περιδικό έλεγχο για το κατά πόσον κρίνεται ε, ένα όχημα ικανό να λειτουργήσει ή όχι να... Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που θα μας απασχολήσει σε περίπτωση που υπάρχει νοθεία στους μετρητές χιλιομετρικών αποστάσεων αυτό συνεπάγεται πάντα μεγάλες κυρώσεις. Αλλά αυτό δεν μας εγγυάται ότι θα πατάξουμε τη συμπεριφορά αυτή. Δηλαδή, αν υπήρχαν πληροφορίες ένα καλύτερο τρόπο να πατάξουμε τι ε, τακτικέ αυτέ και τι πρακτικέ αυτές είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει επιτυχής ε, νοθεία των ε, οδομετρητών. Δηλαδή, κανείς δεν θα ήθελε να δώσει χρήματα σε κάποιον για να αλλάξει τα στοιχεία του οδομετρητή σε περίπτωση που ήξερε ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου των χιλιόμετρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά θέματα ευθύνη, ε, συμφωνώ αλλά τελικά δεν είναι ο κάτοχος του αυτοκινήτου αυτός που προκαλεί το ατύχημα, αλλά ο οδηγός του οχήματος. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να καταλαβαίνω πάντως τι λέτε. ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 21 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι Στις 11 και 25 Απριλίου θα έχουμε την εξέταση και την, της τροπολογίας την ψηφοφορία στην Ήτρε μάλλον και μετά τον Ιούλιο στην Ολομέλεια. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, συνάδελφος Τόγια. Παρακαλώ. Ε, Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά παρουσιάζω αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας που που υποβάλλεται βάσει των περιορισμών που υπάρχουν σε τέτοιου διαδικασίε. Οπότε παραμένει μόνο στα βασικά στοιχεία. Ε, όμως, ε, το, με τη δική μου τη συμβολή όπως και των συναδέλφων θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε το κείμενο και να υπάρχει και η ποικιλία που αρμόζει σε ένα τέτοιο αντικείμενο μελέτης. Στον τομέα αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή από την πλευρά των θεσμικών οργάνων και ιδιαιτέρως από τη δική μας την Επιτροπή. Να θυμίσω το ιστορικό της πρότασης αυτής. Ψήφισμα που εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από το Κοινοβούλιο, τουλάχιστον με συντριπτική πλειοψηφία, στην αρχή της θητείας, Κάτι που ξεκίνησε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς έκθεση για την οποία και εγώ υπήρξα συγγετρία στο Κοινοβούλιο και ασχολείται με τις κοινωνικές ανάγκες καθώς και την κοινωνική οικονομία. Όχι μόνο τις συνεταιρισμούς, αλλά τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τις μη κερδοσκοπικές ενώσεις, τις αλληλασφαλιστικές εταιρείε και όλες όλους τους παράγοντες αυτές που αφορούν την οικονομία, τον ε, κόσμο της οικονομίας, την πραγματικότητα της παραγωγής, την κοινωνική πρόνοια και την απασχόληση. Όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν εταιρείε και επιχειρήσεις κάπως ιδιαίτερες, με συγκεκριμένους σκοπούς. Σκοπό που έχουν, ε, σκοπούς που έχουν να κάνουν με το να δώσουν εργασία, να απασχολήσουν τους πολίτες και ένα στοιχείο αλληλεγγύης, αμοιβαιότητας. Εδώ λοιπόν προσπαθήσαμε να συμβιβάσουμε το στοιχείο της ε, αλληλεγγύης με την οικονομική δραστηριότητα μιας κλασικής επιχείρησης. Γίνεται λοιπόν αυτό το επιχειρήν και το κέρδος είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί και στη βάση επιχειρήσεων με κοινωνική φυσιογνωμία έκθεση αυτή νομίζω ότι μπορεί να κάνει περήφανο το Κοινοβούλιο γιατί μετά ακολούθησαν πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Μπαρνιέ που εγκρίθηκαν και από το Κοινοβούλιο όπως το κοινωνικό επιχειρήν ή διατάξεις που αφορούν ακριβώς με τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική πρόνοια και αυτά βάσει προτάσεων του Επιτρόπου Μπαρνιέ. Ξεκίνησε λοιπόν εδώ ένα νέο ρεύμα, διότι για την κοινωνική οικονομία γινόταν λόγο και γίνεται ακόμα, αλλά σε σχέση με συγκεκριμένε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγα πράγματα γίνονταν. Το ίδιο και για το Κοινοβούλιο. Η έκθεση αυτή λοιπόν έχει πιο συγκεκριμένο αντικείμενο που αφορά τι αρμοδιότητες τη δική μα επιτροπή, αλλά εδώ ε, ε, φυστά την προσοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τι προτάσει που θα ακολουθήσουν. Θα μπορούσαν εδώ να θεωρηθούν αυτά ω ενδείξει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι συγκεκριμένα θα μπορούσε να γίνει, όπω έλεγε και η προηγούμενη έκθεση. Δίνεται έμφαση λοιπόν σε συγκεκριμένα στοιχεία και ζητώ από του συναδέλφου με τι τροπολογίε του να μας βοηθήσουν να είμαστε φάνταστοι. Να πούμε και να σκεφτούμε τι εργαλεία χρειάζονται αυτοί οι συνεταιρισμοί και τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πεδίο ενδιαφέροντος αυτής της έκθεσης αφορά ακριβώς τους συνεταιρισμούς, τις συνεταιριστικέ επιχειρήσεις. Το ρόλο που διαδραματίζουν μάλιστα αυτές κατά τις βιομηχανικέ κρίσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένο το αντικείμενο της έκθεσης. Μιλάμε για συνεταιρισμού βιομηχανικού που προσφέρουν υπηρεσίες, παράγουν δηλαδή, όχι συνεταιρισμού κοινωνικού χαρακτήρα, που αντικείμενο τους είναι το κοινωνικό επιχειρήν, αλλά αντικείμενο του είναι η παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών, και θέλουμε να δούμε τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν στην περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική κρίση παραγωγή. Είναι ευκαιρία αυτέ οι συγκυρίε ή πρόβλημα. Η ευκαιρία που προκύπτει το δείχνει και ο μεγάλο αριθμό συνεταιρισμών. Δεν θα θέλω να δώσω εδώ συγκεκριμένα δεδομένα, διότι αυτά αναφέρονται και στην ε, πρόταση ψηφίσματο. Όμω οι συνεταιρισμοί που παράγουν ε, αγαθά και υπηρεσίε, βιομηχανικοί, είναι το 5% του ΑΕΠ αυτό δείχνει μια πραγματικότητα που δεν είναι τα ευκαταφρόνητη. Και αυτό μας συμφέρει να εξεταστεί για δύο λόγους. Πρώτον, διότι και αυτοί οι συνεταιρισμοί, όπως και άλλοι, με άλλου είδους προϊόντα κοινωνικού χαρακτήρα, αυτοί λοιπόν οι συνεταιρισμοί παρέμειναν και άντεξαν καθόλου την περίοδο της κρίσης. Τα δεδομένα μας έδειξαν ότι η απασχόληση παρέμεινε στα ίδια ποσοστά, ο όγκος παραγωγής αυτών των ε, συνεταιρισμών παρέμεινε στα... αυξήθηκε και Μιλάμε για συνεταιρισμού που και κατά τη διάρκεια της κρίσης μπόρεσαν να αντισταθούν στους ανέμους ε, αυτούς, τους θυελώδεις. Και η κοινωνική τους επιχειρηματικότητα τους ε, έκανε και πιο ανθεκτικούς. Εδώ στο σκοπό γενικότερα έχουμε να αυξήσουμε την απασχόληση παρά να απολύσουμε ανθρώπους. Όμως υπάρχει κι άλλο ένα δεδομένο που φαίνεται από τις μελέτες. Μία μελέτη που αναφέρει λόγου χάρη ότι ακόμα και στην περίοδο της κρίσης προκύπτουν νέοι συνεταιρισμοί. Όχι μόνο αντέχουν λοιπόν και αντίστανται, αλλά το ποσοστό ε, ανάπτυξης τους ε, βελτιώνεται τη στιγμή, ε, σε στιγμές κρίσης παρά σε στιγμές άνθησης της οικονομίας. Αυτό δείχνει τι γίνεται με ε, επιχειρήσεις νέων ή γυναικών. Δηλαδή κάποιες φορές αυτό που τους οδηγεί να διακινδυνεύσουν και να επιχειρήσουν τους νέους και τις γυναίκες δεν είναι μόνο η επιχειρηματικότητά τους και το πνεύμα του επιχειρήν αλλά και οι συγκυρίες δυσχέρειας. Τρίτο στοιχείο τώρα ότι οι συνεταιρισμοί αυτοί μπορούν να αποτελέσουν μια καλή επιλογή μετατροπής μιας θνίσκουσας επιχείρησης ή που ε, αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα διαχείρισης, management δηλαδή. Επιχειρήσεις με καλά προϊόντα, ε, με καλές, με καλούς εργαζομένους και αξιόλογους εργαζομένους, αλλά λόγω κρίσης αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες. προκειμένου λοιπόν να μην πτωχεύσουν, μπορούν να επενδύσουν σε μια τέτοιου είδους επιχειρηματική δράση. Τέτοια δεδομένα βλέπουμε και στην Ιταλία, στη χώρα μου, αλλά και στη Γερμανία και τη Γαλλία. Και ανακάλυψα με μεγάλη έκπληξη ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή της Δανίας ή άλλων χωρών έκπληξη διότι δεν ήμουν γνώστρια, όχι γιατί δεν το γνώριζαν οι υπόλοιποι, εγώ δεν το γνώριζα. Πάντως έκπληξη διότι και εδώ οι συνεταιρισμοί ταυτόχρονα με άλλες μορφές όπως ανάκτησης από το management του επιχειρηματικού κεφαλαίου και των ε, υπόλοιπων συνεταίρων ε, ή των εργαζομένων, αυτό ίσως να είναι μια επιλογή για να αποφύγει κανείς την πτώχευση. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικός αριθμός περιπτώσεων που δείχνουν ότι αυτή είναι μια πιθανή λύση. Παρ' όλα αυτά, καθώς το κοινοβούλιο μας στο πλαίσιο της επανεκβιομηχάνησης ε, θεωρεί ότι η καλύτερη επιλογή είναι να γίνονται αναδιαρθρώσεις στα επίπεδο των επιχειρήσεων, αυτό τι η περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να προκαλέσει όλο μας το ενδιαφέρον και την προσοχή. Νομίζω λίγη χρόνο μου, σωστά. Όχι, ναι. Ξεχάσαμε το χρόνο. Ε, δυόμιση λεπτά παραπάνω. Δύο λεπτάκια μόνο και για τον τίτλο. Να εξηγήσω τη σημασία του θέματος αυτού με τηλεγραφικές παρατηρήσεις. Το πιο σημαντικό είναι το τι θα κάνουμε τι πρέπει να γίνει. Ε, θα μπορούσαν να υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία ad hoc με άλλε μορφέ στήριξη. Εδώ η Ευρώπη θα μπορούσε να προβλέψει μια δημοσιονομική γραμμή ή ένα πιλωτικό σχέδιο, αλλά πραγματικά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να διασφαλίσουμε το κεφάλαιο, να προστατεύσουμε το απαραίτητο κεφάλαιο για τέτοιου είδου ε, επιχειρηματικέ πρωτοβουλίε. Αυτό λοιπόν μα ενδιαφέρει. Τι θα πρέπει να γίνει. Και προ αυτή την κατεύθυνση θα θέλαμε να κινηθούν και οι τροπολογίε για να εμβαθυνθεί περισσότερο αυτό το δεύτερο τμήμα τη έκθεση. Πρόεδρο, ευχαριστώ την κυρία Τόγια, ο κύριο Καντζάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω τα όσα είπε η Πατρίτσια, ιδιαίτερο αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, τη συγκυρία της κρίσης, είναι θετικά. Πραγματικά θα πρέπει το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας, να δώσει προσοχή σε αυτό το θέμα. Σέβομαι τα όσα ακούστηκαν, αλλά θα ήθελα να επιστήσω εδώ και την προσοχή μας σε κάτι. Να προσέξουμε λίγο. Κάποιες διευκολύνσεις ε, υπέρ των οποίων θα μπορούσα να ταχθώ για να δοθεί κίνητρο να συνενώσουμε εδώ και την επιχειρηματική δραστηριότητα με τις ανάγκες απασχόλησης αυτό είναι κάτι που το θέλουμε σήμερα, ιδιαίτερο σήμερα. Ιδιαίτερο στις προσεχείς ημέρες, την επόμενη ακόλουθη περίοδο με τις προοπτικές που υπάρχουν. Μην το ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει και ένα παρελθόν και θα πρέπει να φροντίσουμε το σύστημα διευκολύνσεων να μην διαταράξει τους κανόνες βάσει των οποίων λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Φοβούμε ότι εδώ μπορεί να υπάρχουν ε, κάποιες περιπτώσεις συνεταιριστική δράσης και κοινωνικών επιχειρήσεων που μπορεί να συγκαλύπτουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό δεν είναι απλός φόβος, διότι τέτοιες περιπτώσεις τις είδαμε και στο παρελθόν. Βεβαίως, αυτό δεν θα πρέπει να μειώσει τη θετική αποτίμηση από πολιτική σκοπιά αυτή τη δραστηριότητα. Πάντως, ευελιξία, η ευελιξία και η μακρά παράδοση που έχουμε δει να επικεντρώνονται και να, παρατηρούνται σε αυτό το σύστημα των συνεταιρισμών είναι μια καλή επιλογή για να αποφύγουμε προβλήματα και τραυματισμούς στο μέλλον ως προς τους συνεταιρισμούς αυτούς. Επι, επαναλαμβάνω ότι η συνένωση επιχειρηματικής δράσης και εργασίας είναι αποτέλεσμα, είναι καρπός κοινωνικού συνεταιρισμού, ε, συνεταιριστικής δράσης, όπως παρατηρεί και το έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας. Να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό και να προσπαθήσουμε από κοινού όλοι να προσφέρουμε μια θετική συνεισφορά ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα που να δώσει αποκρίσεις και απαντήσεις σε τόσες επιχειρήσεις που σήμερα ζουν στιγμές ακραίων δυσχεριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Καντσάν. Ο συνάδελφος Πρόντε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Πατρίτσια Τόια Εδώ συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα, διότι περνάμε μια στιγμή όπου εν τέλει υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για, και ευαισθησία για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Βλέπουμε επιχειρήσεις, επιχειρήσεις προσώπων και αυτό μας ενδιαφέρει πλέον και όχι οι επιχειρήσεις κεφαλαίων. Πρέπει να είμαστε σε θέση αυτή την ευαισθησία μας να την αποδείξουμε και έμπρακτα. Διότι ε, θέλουμε να δείξουμε ακριβώς ότι μας ενδιαφέρει το κοινό ε, συμφέρον, το καλό της ε, κοινωνίας μας. Υπάρχει μια δυναμία εδώ στην, στις επιχειρήσεις βέβαια αυτές, η κεφαλαιοποίησή τους. Θα πρέπει καταρχάς να, να υπάρξει ανάληψη ευθυνών από τις ενώσεις συνεταιριστικών επιχειρήσεων διότι υπάρχει σύγκληση από πολλές ε, ενώσεις που δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα στην Ιταλία βάσει πολιτικών ε, προδιαγραφών και οι οποίες τώρα ενοποιούνται. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα αυτές οι ενώσεις οι ίδιες να αναλάβουν ευθύνες ώστε όλες οι ανάλογες επιχειρήσεις να είναι αντικείμενο διαχείρισης που να συμμορφώνεται απολύτως με τις γενικές ε, αυτές αρχές. Για την κοινωνική λοιπόν ευθύνη των επιχειρήσεων, κάτι που θεσμικός ε, γίνεται μια ε, επιταγή, θα πρέπει αυτό να διαμορφωθεί ως ένα ωφέλιμο στοιχείο για ολόκληρη την κοινωνία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τώρα ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κάποιος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Ιωακιμίδης, είμαι στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και εκεί έχουμε μία μονάδα η οποία ασχολείται με την κοινωνική οικονομία και πιο συγκεκριμένα με τους συνεταιρισμούς. Και αυτό εδώ και πάνω από 20 χρόνια τώρα. Τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια εμείς πιστεύουμε ότι αναπτύξαμε μία πολιτική η οποία τη σήμερα ημέρα διασφαλίζει στους συνεταιρισμούς δίκαιους κανόνες όταν συγκρίνονται με τις άλλες τις κεφαλαϊκές επιχειρήσεις. Η έκθεση τώρα της κυρίας Τόγια συμπεριλαμβάνει όλους τους τομείς όπου μπορεί ακόμα να υπάρχει περιθώριο για προτάσεις και νέες ιδέες. Εμείς αντιλαμβανόμεθα ότι απευθύνεται κυρίως στα κράτη-μέλη και εννοείται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει με την εφαρμογή τέτοιων μέτρων. Διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να μας στηρίξει ηθικά στην εφαρμογή των μέτρων αυτών και εμείς ευχαρίστως να συνεργαστούμε με την κυρία Τόγια όσον αφορά τις διάφορες ιδέες της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπενθυμίζω ότι η κατάθεση... Α, δεν τελειώσαμε. Συγγνώμη, συγγνώμη, κάτι ξέχασα. Το λόγο έχει βέβαια η συνάδελφος η κυρία Τόγια. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, όχι μόνο όσους εκφράστηκαν σήμερα, αλλά και όσοι από τη θέση του σκιώδου συγκητού ή οποιαδήποτε άλλη θέση θα συμβάλλουν στην αμπλουτισμό της έκθεσης αυτής που το έχει ανάγκη, γιατί το επιβάλλει και το ίδιο το θέμα της έκθεσης. Θα το ζητούσαμε αυτό και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εργαστούμε παραλληλό και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσουν αυτές τις δομές που κάνουν ό,τι μπορούν ε, τη σύμπρονη μέρα, αλλά θα πρέπει να δυναμωθούν για να προωθήσουν και τη μηχανική πολιτική και την πολιτική των επιχειρήσεων. Είναι τόσε πολλέ. Είναι μια συμβολή που θα πρέπει να τη δώσουμε λόγω τη μορφή που έχει πάρει η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, αλλά και για του σκοπού τη εργασία και τη απασχόληση. Θα εργαστούμε λοιπόν ε, μαζί και θα είμαστε και απαιτητικοί. Ε, απαιτητικοί με τι προτάσει που θα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βεβαίω. Πρόεδρο. Ευχαριστούμε. Κλείνουμε και με το σημείο αυτό. Να θυμίσω ότι η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών είναι 25 Μαρτίου το μεσημέρι. Θα συζητηθεί στην Ήτρε στις 25 Απριλίου και στην Ολομέλεια μάλλον τον Ιούνιο του 2013. Ωραία, το ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και τώρα βάσει του άρθρου 70, εδάφιο 4 του εσωτερικού κανονισμού, έχουμε μια ενημέρωση σχετικά με τους ανεξελίξει τριμερούς διαλόγους. Κατά πρώτον, να δώσω τον λόγο στον κύριο Κρόιτσμαν για πέντε λεπτά για να μας ε, παρουσιάσετε πώς έχει κατάσταση. Ναι. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στις 29 Ιανουαρίου 2013 έγινε τρεμερής διάλογος και συζητήσαμε διάφορα θέματα για την κατανομή των ε, πόρων του προπολογισμού. 60% πρότεινε το Κοινοβούλιο, 55% το Συμβούλιο. Η διαφορά φαίνεται να μην είναι τόσο μεγάλη και θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Ένα άλλο θέμα ήταν το θέμα του διοικητικού άχθους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να επικεντρωθεί σε θέματα διοικητικού άχθους, ενώ το Συμβούλιο το έχει επεκτείνει σε ρυθμιστικό άχθος, διοικητικό και ρυθμιστικό άχθος. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τον νομοθέτη. Και τώρα συζητάμε κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δύο όροι. Administrative and regulatory burden. Το θέμα του, των τιμών ορίου και του ορίζοντα 2020 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα συνάδει με το αποτέλεσμα που περιλαμβάνεται στον ορίζον 2020. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να καταφέρουμε ένα ταχύ αποτέλεσμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ανησυχία γιατί ενδεχομένως να υπάρχει αλληλεπικάλυψη με το πρόγραμμα του ορίζοντας 2020 και αυτό θα αυξήσει το διοικητικό σε τροπολογία και πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Συμφωνήσαμε ότι είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό και θα πρέπει να επιληθεί σε πολιτικό επίπεδο. Συγκεκριμένη ομάδα στόχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο, διέγραψε τις σχετικές αναφορές στο, στην αιτηλογική ε, σκέψη 11 για τον τουρισμό. Υπάρχει ευρεία συμφωνία σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και συμφωνήθηκε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων δεν ήταν τόσο σημαντικές. Εφαρμόσαμε, μάλλον υπήρξε μια τεχνική ομάδα η οποία συνεχίζει τις εργασίες της και ο επόμενος τριμερής διάλογος προγραμματίζεται για της 9 Απριλίου του 2013 το πρόβλημα είναι κατά πόσον θα έχει ολοκληρωθεί η εργασία. Γιατί μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά το έργο της ε, τεχνικής ομάδας. Αυτά λοιπόν για την κόσμο. Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Κρόισμαν για τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε και τώρα ο κύριος Γκλάντε που καθόταν κύριο Κάλφιν, Κάλφιν μάλλον, συγγνώμη, και θα μας εναμερώσει για τη χρήση των πληροφοριών στο δημόσιο τομέα. Σας ευχαριστώ. Αντικαθιστώ σήμερα πολλού ε, συναδέλφου, αλλά είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση. Εξ ονόματο λοιπόν τώρα του συναδέλφου να πω ότι οι τριμερεί διάλογοι ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο μετά την ε, ε, έγκριση της ε, έκθεσης στην Επιτροπή. Έγινε κάποια ανταλλαγή απόψεων με την Κυπριακή Προεδρία και την σχετική αρμόδια Γενική Διεύθυνση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 17 Ιανουαρίου και 18 Φεβρουαρίου έγιναν συναντήσεις στα πλαίσια του τρομερούς διαλόγου. Για τις 25 Μαΐου προγραμματίζεται η επόμενη συνάντηση και σκοπός θα είναι να πετύχουμε πολιτική συμφωνία για την πλειοψηφία των σημείων. Έχουμε το άρθρο 6 για το ρόλο και το ε, άρθρο 4 για το ρόλο των ε, αμερόληπτων σωμάτων και το ε, άρθρο 11 η άποψη του Κοινοβουλίου